Επίση επίσης μου ανακοίνωσε ότι έχει προσχωρήσει στην ομάδα των Πρασίνων. Οι αρμόδιες αρχές της Ουγγαρίας μου ανακοίνωσαν την εκλογή του κυρίου Ερικ, του κυρίου Μπάνκι, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Ζάνο Σάντερ, ο οποίος εξελέγει στην Ευρωτερική Βουλή και θα ήθελα να υπενθυμίσω τη δυνάμη του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού. Όσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι εξουσίες τους συμμετέχουν στα συνεδριάσεις και τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εφόσον βεβαίω δεν υπάρχει συμβατότητα ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων του Βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, έχει καταθέσει ο κύριος Μπάνκι δήλωση γραπτή η οποία εξηγεί ότι δεν υπάρχει συμβατότητα με τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλώ ήρθατε λοιπόν. Η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων στη συνεδρίαση της 30 η Μαΐου του 2012 επιβεβαίωσε τις εντολές ε, των βουλευτών από 18